Euh, Ευχαριστώ για την πειθαρχία σας και την προσοχή σας. Από ό,τι κατάλαβα, ο Ζαν Κρός μου το λέει, αυτό είναι μεγάλη πρεμιέρα. Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωκοινοβουλίου και Επιτροπή ε, της Επιτροπής των Περιφερειών βρίσκεται εδώ για να συζητήσουμε σημαντικά θέματα. Για να συζητήσουμε την Ήπεθρο ε, και την πολιτική, τη μελλοντική για την ανάπτυξη Πέθρου. Κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Σιγητά, αγαπητοί συνάδελφοι της Επιτροπής ε, Γεωργίας και τη Επιτροπή ΝΑΤ, τη Επιτροπή των Περιφερειών, είναι χαρά και τιμή ειλικρινή χαρά για μένα που καλωσορίζω τους συναδέλφους της Επιτροπής ΝΑΤ, της Επιτροπής των Περιφερειών. Η συμμετοχή του στην ανταλλαγή απόψεων, η σημερινή ανταλλαγή απόψεων για τη μελλοντική πολιτική ανάπτυξη της υπαίθρου Θεωρώ ότι μόνο ότι εντάσσεται με φυσικό τρόπο στο πλαίσιο των θεσμικών σχέσεων που θέλουμε να ενισχύσουμε, αλλά και είναι ιδιαίτερος ε, επίκαιρη. Υπάρχουν προσδοκίες από πλευράς των περιοχών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και θα γίνει αξιολόγηση των πολιτικών και θα διαμορφωθούν οι μελλοντικέ πολιτικές στο μέσα ο κ. Πρόεδρος κ. Σικέρσκι, που θα καταφτάσει αργότερα, σήμερα το απόγευμα, ήδη δύο φορές είχε τη δυνατότητα να μιλήσει και να μιλήσει στην Επιτροπή ΝΑΤ και να εκτιμήσει τη σοβαρότητα και τη ζωτικότητα της συζητήσεως που διεξήχθηκε. Είμαι σίγουρος ότι οι σημερινές ανταλλαγές απόψεων, οι σημερινές μας συνομιλίες θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο επιτροπές μας θα εμπλουτιστούν αμοιβαία από την ποικιλομορφία των απόψεων και από τις κοινέ ανησυχίε που θα εκφραστούν. Το διακύβευμα της υπαίθρου είναι και το μελλοντικό διακύβευμα εν ώψη της μελλοντική μεταρρυθμίσεως του τομέα. Άρα όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να ρίξουμε μια ματιά αντικειμενική μέλλοντος στραφή διότι υπάρχουν αλλαγές επιταχυνόμενες και η γίνεται αυριανός στόχος για μας που είμαστε υπεύθυνοι. Να σας πω λοιπόν πώς θα εργαστούμε. Να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής ΝΑΤ, τον κύριο Αντώνη Ζεράρ Μπουκάναν, ο οποίος θα εκφράσει την άποψη τη τοπική της τοπικής αυτοδιοίκησης για το μέλλον της πολιτικής για την Ήπεθρο. Μετά ο κ. Ράντερ Λάντ θα πάρει το λόγο, ο εισηγητή θα παρουσιάσει το περιεχόμενο τη Λευκή Βίβλου για την πολιτική για την Ήπεθρο. Οι δύο παρεμβαίνοντε και είμαστε αυστηροί στο χρόνο. Εδώ θα πρέπει, λέγω, οι δύο παρεμβαίνοντε να, να μιλήσουν για ένα τέταρτο ο καθένα. Μετά θα δώσουμε το λόγο για ένα δίλεπτο στον καθένα, στους συντονιστές των δύο επιτροπών μας θα ξεκινήσουμε από τους συντονιστές της Επιτροπής ΝΑΤ και έτσι θα ακούσουμε με τη σειρά τον κύριο Πέτερσεν, τον κύριο Ζεμπλεουίξ, τον κύριο Κάινεν, τον κύριο Στένσον και τον κύριο Χάτς με την προναφερθή σας σειρά. Και μετά θα ακουστούν οι συντονιστές της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σύμφωνα με την σειρά που μιλούν οι πολιτικές ομάδες, πασίγνωστη σειρά που ακολουθείτε. Στον υπόλοιπο χρόνο θα υπάρξει γενικότερη συζήτηση. Θα συμμετάσχουν οι παρόντες σύμφωνα με την αρχή προσέλκυσης προσοχής του Προέδρου. Και μετά θα συνοψίσουμε τις απόψεις θα είναι πλούσιες οι ανταλλαγές απόψεων. Θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια φωτογραφία της απόψεως που έχουμε διαμορφώσει και για τις κοινέ προσπάθειες. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Αντώνη Ζεράρ Μπουκάνων για να μας μιλήσει από πλευράς τοπικής αυτοδιοίκησης και πώς βλέπουν οι αρχές αυτές το μέλλον της ε, πολιτικής για την ανάπτυξη της Πέτρου. Thank ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Νιώθω μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ, σε αυτή την ε, πρώτη κοινή διάσκεψη με την ε, Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω αυτή η πρώτη κοινή διάσκεψη να αποτελέσει την ε, απαρχή στενότερης συνεργασίας για τα δύο θεσμικά όργανα. Θα ήθελα να σας μεταφέρω την ε, συγγνώμη της ε, Προέδρου της Επιτροπής ΝΑΤ, της Φρανσίνα Αρμενγκόλη Οσίας, που δυστυχώς κολλείεται σήμερα. Ένιωσε μεγάλη απογοήτευση λόγω της απουσίας αυτής, γιατί η εξασφάλιση αναγνώρισης ε, των αγροτικών ζωνών ως κομβικό σημείο για την ανάπτυξη και την καινοτομία που μπορούν να συμβάνουν στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική του 2020 είναι τμήμα των ισορροπημένων σχέσεων με τις αστικές περιοχές και η αναγνώριση αυτή αποτελεί η πρωταρχική προτεραιότητα της Επιτροπής ΝΑΤ, της Επιτροπής Περιφερειών. Ονομάζομαι Τζόνι Μπουκιάνα και ε, είμαι από ένα δημοτικό συμβούλιο της ε, Σκωτίας και ε, είμαι αντιπρόεδρος της ΝΑΤ, της Επιτροπής ΝΑΤ. Η περιφέρειά μου, το Ιστρέτρεσερ, είναι κοντά στην Γλασκόβη και έχει 92.000 τοπικό πληθυσμό, 1,7% του συνολικού σκοτσέζικου πληθυσμού. Επίσης, έχουμε 17.400 ε, εκτάρια, 75% εκ των οποίων αποτελούν αγροτικοί ε, αγροτικές ζώνες. Και ευχαριστώ θερμά τον κύριο Σικέσκη που ήρθε στην Επιτροπή, συνεδρία της Επιτροπής ΝΑΤΟ Μάρτιο για να συζητήσουμε από κοινού το μέλλον της ε, ε, Αναπτυξιακή πολιτική τη Υπέθρου σε συνεργασία με του τοπικού και περιφερειακού ε, εκπροσώπους. Και ήταν, αυτό ήταν το αναρκτήριο λάκτισμα για την, ε, και για τη σημερινή μας συνάντηση. Και είμαι ιδιαίτερα ευγνώμων στα μέλη της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έλαβαν μέρος στο σεμινάριο για το μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής στην Υπέθρο για την προγραμματική περίοδο του 2020 που έγινε 19 Σεπτεμβρίου σε συνεργασία με την Διεθνή Ένωση για την Αγροτικότητα, το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη και τη διακομματική ομάδα ΡΑΜΡΑ για τι αγροτικέ ορεινέ και εξόχω απόγευτε περιοχέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μάλιστα η υποστήριξη που, που έδειξαν στο σεμινάριο ενίσχυσε την ε, δέσμευσή μας υπέρ της ε, προώθησης ε, της προσπάθειας αυτής για να συμπεριληφθεί η ανάπτυξη της υπαίθρου στην στρατηγική του 2020 και μάλιστα σε νέα ε, Νοεμβρίου είχαμε μια κοινή συνεδρίαση με την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή για να εορτάσουμε την 20η επέτειο της πρώτης διάσκεψης του ΚΟΡΠ που σηματοδότησε τα γεννητούρια ούτως υπήν της ε, αγορετικής αναπτυξιακής πολιτικής. Και μάλιστα ε, φάνηκε και με την παρουσία του κ. Σεκέσκη στις συζητήσεις με τους τοπικούς και περιφερειακούς ερετούς ότι ε, η κοινωνία των πολιτών και η ΟΤΑ έχουν κοινέ ανησυχίε ε, και ζητούν κοινέ δεσμεύσει ε, για την αναγνώριση των ε, αγροτικών ζωνών, που θα πρέπει να αναγνωριστούν ως κομβικά σημεία για, την, τον εξυγχρονισμό και την καινοτομία και θα πρέπει να συμπεριληφθούν στη στρατηγική του 2020 στα πλαίσια ενός μιας ισορροπημένης σχέσης. Αυτή είναι η βασική προτεραιότητα της Επιτροπής ΝΑΤ. Και μάλιστα η δεύτερη διάσκεψη του ΚΟΡΚ του Σεπτεμβρίου έδειξε μια ε, πλέον έμφαση στο θέμα της ανάπτυξης της υπαίθρου. Και εναπόκειται τώρα σε εμά να συνεργαστούμε στενά ώστε να συμπεριληφθούν αυτά τα συμπεράσματα και να εφαρμοστούν σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Και μάλιστα με την ε, γνωμοδότησή μας ε, για την καινοτομία και την, τον εξυγχρονισμό της γεωργικής οικονομίας του κ. Ράντελ Λάντς, η Επιτροπή μας ε, απευθύνω μια έκκληση προς το κίνημα για την Ευρωπαϊκή Υπεθρό και τη διακομματική ομάδα Ρούμπρα για, για μια λευκή βίβλο για την αγροτικότητα που θα αποτελέσει το σημείο εκκίνησης για την αναπτυξιακή αγροτική πολιτική μετά το 2020. Και μάλιστα ο κ. Λάντς αργότερα θα σας παρουσιάσει τις πρακτικές προτάσεις και συστάσεις της γνωμοδότησής του. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω την ανάγκη, την επιτακτική ανάγκη που συνιστά η σύνταξη μιας λευκής βίβλου για την αγροτικότητα και ευελπιστώ ότι η Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα μας στηρίξει σε αυτό το αίτημα. Οι αγροτικές και διάμεσες ζώνες αποτελούν το 91% της ευρωπαϊκής επικράτειας, 60% του πληθυσμού της και παράγουν 43% τη ακαθάριστη της αξία. προστιθέμενης αξίας. Ε, ε, παρέχουν το 56% των θέσεων εργασία. Παρ' όλα αυτά, οι αγροτικέ ζώνες υστερούν σε σχέση με τι αστικέ. Ε, ο μέσο όρο του ΑΕΠ στι αγροτικές ζώνε είναι 73% χαμηλότερο από ό,τι στι αστικέ. Και η διαφορά αυτή είναι ιδιαίτερα ορατή στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού διαμένει στην Ήπεθρο, στι αγροτικέ ζώνε. Έχουμε μια πληθώρα λοιπόν προκλήσεων και βλέπουμε ότι οι αγροτικές ζώνες υστερούν σε σχέση με τις ε, αστικές. Οι δημογραφικέ προκλήσει είναι από τα κομβικά σημεία της κοινή γεωργικής πολιτικής. Ο αριθμό των ε, γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρώπη μειώθηκε κατά 20% από το 2007 μέχρι το 2013 και από 13,6 εκατομμύρια πέρασε 10,8 εκατομμύρια μέσα σε μία εξαετία με βάση τα τελευταία επίσημα στατιστικά στοιχεία της Eurostat. Γνωρίζω ότι η, Επιτροπή Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμμερίζεται αυτές ε, τις ε, παρατηρήσεις ε, και φάνηκε στην πρόσφατη έκθεση του Ερίκ Θα πρέπει λοιπόν να, να αναβαθμίσουμε την κάπως δημόσια πολιτική που θα ωφελεί τους πάντες, θα λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικές ανάγκες και θα αντιμετωπίζει και τις προκλήσεις στην απασχόληση. Επίσης, η ανανέωση των γενεών είναι ε, ανερχόμενο πρόβλημα. 30% των διαχειριστών γερικών εγκαταλέψεων είναι άνω των 65 ετών. Και ελάχιστοι είναι οι, οι νέοι ε, γεωργοί, γιατί θεωρούν δύσκολο το να ξεκινήσουν μια γεωργική δραστηριότητα που θα τους εξασφαλίζει ένα αξιοπρεπές εισόδημα. Γενικώ, οι χαμηλές ε, αμοιβές, τα χαμηλά εισοδήματα των αγροτικών δραστηριοτήτων ε, σε σχέση με τις υπόλοιπους ε, κλάδους οικονομίας είναι πολύ απογοητευτική και αποθαρρυντική. Και μάλιστα στο Φεβρουάριο στην, ε, ε, στην Ολομέλεια θα ασχοληθούμε με το θέμα αυτό. Υπάρχει κρίση που έχει πλήξει ιδιαίτερα τον αγροτικό τομέα. Οπότε γι' αυτό οι υπεθρώσεις ζώνες δεν είναι ιδιαίτερα ελκυστικές για διαβίωση γιατί δεν προσφέρουν ούτε επαρκή παιδεία, ούτε αρκετές υπηρεσίες πολιτιστικέ, κοινωνικές και ε, υγείας. Ε, μικρή προσβασιμότητα, μεγαλύτερε αποστάσεις από, από τα κέντρα λήψη αποφάσεων και από τα, τους ερευνητικούς κόμβους. Υπάρχει το τεχνολογικό χάσμα, γι' αυτό και θα πρέπει να διεκδικήσουμε επέκταση της ευρυζωνικότητας ε, των τηλεπικοινωνιών. Οι δεμοί θα εξακολουθούν να υστερούν οι αγροτικές ζώνες και μάλιστα το 2003 μόνο το 25% των ε, αγροτικών ζωνών είχαν ε, ευρυζωνικό ίντερνετ ε, σε σχέση με το 68% και 90% των οικοκυριών που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ είναι σε αγροτικές ζώνες. Και ενώ η έννοια, η ιδέα της έξυπνης πόλης έχει γίνει η πρωταρχική επιλογή των πολιτικών εθνών για τις μελλοντικές προκλήσεις, η Επιτροπή Περιφερειών θεωρεί ότι αντίθετα θα ήταν αδύνατο να υλοποιήσουμε τους στόχους ανάπτυξης και ε, απασχόλησης αν δεν ενισχύσουμε την εδαφική συνοχή στην Ευρώπη και χωρίς να αξιοποιήσουμε όλες τις πηγές του δυναμικού της ανάπτυξης συμπεριλαμβανομένων και των αγροτικών ζωνών. Και μάλιστα οι προετοιμασίες για την περίοδο προγραμματισμού μετά το 2020 έχουν ξεκινήσει ήδη. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε εμπεριστατωμένη συζήτηση για τις ανάγκες της υπαίθρου των αγροτικών ζωνών, ώστε η πολιτική μετά το 2020 να είναι σημαντική και για τις αγροτικές ζώνες και να έχει και προστιθέμενη αξία και η συμβολή σε, ένα, μια ευφύ βιώσιμη και ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμού που είναι ο στόχος στρατηγικής του 2020, ε, υποαξιοποιείται προς το παρόν. Γι' αυτό και ενώ ζητούμε τη βοήθειά σας για την ε, Λευκή Βίβλο. Επαναλαμβάνουμε την έκκλησή μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η δεύτερη διάσκεψη του ΚΟΡΠ και η στρατηγική μετά το 2020 θα πρέπει να θεωρηθεί ως ευκαιρία για να ε, θέσουμε ως επίκεντρο τις ανάγκες των αγροτικών ζωνών και να δώσουμε ευκαιρίες σε αυτούς που έχουν επιλέξει αυτές τις περιοχές για την διαβίωση του, τη διαμονή τους. Θα πρέπει λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία, να θετήσουμε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση και να απαντήσουμε στο ερώτημα προς τη γεωργία. Επίσης θα πρέπει να στηρίξουμε την προσπάθεια διαφοροποίησης των αγροτικών ζωνών και επίσης να αντιληφθούμε ποια είναι ε, και με πιο ολοκληρωμένο τρόπο την Ευρωπαϊκή Γεωργική Πολιτική. Όπως λέει και η διάσκεψη και η διακήρυξη CORK 2.0 ε, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την ε, ανάπτυξη με όρους και την ανάπτυξη που θα καταμετράτε σε τοπικό επίπεδο, σε αγροτικό επίπεδο και επίσης να μην μειώσουμε τις επενδύσεις ε, σε υποδομές ε, και στην κρίσιμη μάζα που θα πρέπει να δημιουργήσουμε στην, ε, στις γεωρικές περιοχές και συγκεκριμένοι στόχοι και δεσμεύσεις όπως η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου και η αναζήτηση θέσεων απασχόληση υψηλή ποιότητα είναι βασική μας στόχη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μπουκάνον για αυτά που μας είπατε. Θα δώσουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Βαντερλάντ, για να μας παρουσιάσει το περιεχόμενο της Λευκής Βίβλου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ξεκινήσω επαναλαμβάνοντα αυτά που είπε και ο κύριος Πιουκάναν, ότι όντως χαιρόμαστε που βλέπουμε τη συνέχιση της ε, πολύ επικοδομητική συνεργασία μεταξύ μόνο και της Επιτροπής ε, Άγκρη και της Επιτροπής ΝΑΤ, της Επιτροπής των Περιφερειών. Ε, μου θυμίζει και τις ημέρες που ήμουν Ευρωβουλευτής. Χαίρομαι που ξανάρχομαι. Κυρίες και κύριοι, η Επιτροπή των ε, περιφερειών θεωρεί ότι μόνο με μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στην δημόσια πολιτική θα είναι δυνατόν να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σε κάθε μέρος της Ευρώπης και ειδικότερα στις γεωργικές περιοχές. Πρέπει να επικεντρωθούμε συγκεκριμένα σε τρία θέματα. Πρώτον, το μεγαλύτερο θέμα θα είναι η οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη της θέσης εργασίας και την εδαφική συνοχή. Δεύτερον, η ε, διαφοροποίηση των σημείων εισόδου και η ένταξη της ε, γεωργικής διάστασης της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η συνέχιση της εναρμόνισης ε, των διαρθρωτικών ταμείων και των κανόνων αυτών με το στρατηγικό πλαίσιο. Η Επιτροπή Περιφερειών ομόφωνα ενέκρινε μια γνωμοδότηση ιδίας πρωτοβουλίας για την καινοτομία και την εξυγχρονισμό στην αγροτική οικονομία με μεγάλη μου τιμή υπήρξα ο εισηγητής αυτής της έκθεσης και σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερείς προτάσεις σε αυτούς τους τομείς δράσης. Ξεκινώ λοιπόν με το πρώτο θέμα. Είναι η οικονομική υποστήριξη από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, την απασχόληση και την εδαφική συνοχή. Παρόλο που η εδαφική συνοχή είναι ένας από τους στόχους που ορίζονται στη συνθήκη της Λισαβόνας, είναι κάπως ε, περίεργο αλλά και απογοητευτικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή τα διαρθρωτικά ταμεία όπως λειτουργούν αυξάνουν τις περιφερειακές ε, διαφορές. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις σχετικά με το μέλλον της κοινή ε, γεωργικής πολιτικής και πώς θα της δώσουμε μια βάση νομιμοποίησης. Οι επιχορηγήσεις είναι ο στόχος ε, μεγάλης κριτικής διότι δίνουν μεγαλύτερη, ε, μεγαλύτερο βάρος σε μεγάλες παραγωγικές ε, εκμεταλλεύσεις ε, που είναι πιο εξειδικευμένες και σε συγκεκριμένα συγκεντρωτικά συστήματα. Γεγονός που ενισχύει τις διαφορές και κάνει τις μικρές εκμεταλλεύσεις να εξαφανίζονται. Οι οικονομικές, λοιπόν, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις είναι πράγματα που σας εξήγησε ο κύριος Μπουκάναν, είναι ε, ο λόγος που έχουμε αυτές τις προτάσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης και της ε, ενσωμάτωσης στις ε, αγροτικές περιοχές. Επίσης, η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης, που είναι σημαντική για να αντισταθμιστούν αυτές οι διαφορές, που είναι πρώτος, υπό τον πρώτο πυλώνα της κοινή αγροτικής πολιτικής, δεν μπόρεσε να ανατρέψει τις τάσεις αυτές. Ο κ. Πιουκάναν Επίση, σας έδωσε μια λεπτομερή ανάλυση του προβλήματος ε, στην ακρόαση που έγινε στη Σεπτέμβριο του 2015 και σύμφωνα με τους αρχικούς λοιπόν ε, υπολογισμούς ε, της Κομισιόν, τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης που δίνεται για τη γεωργία με την έκτη προτεραιότητα την προώθηση δηλαδή της κοινωνικής ένταξης, τη μείωση της φτώχειας και την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές λαμβάνει μόλις 15% του συνολικού προϋπολογισμού. Η συγχρηματοδότηση ε, των μέτρων, ε, λοιπόν, ε, αποτελεί πρόβλημα για τις περιφέρειες με, λιγότερες, με λιγότερους πόρους. Και αυτό εξηγεί και τη λιγότερη απορρόφηση των πόρων από κάποια κράτη-μέλη. Δυστυχώς, τα νούμερα επιβεβαιώνουν τις ανησυχίες της, της Επιτροπής των Περιφοριών για τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών. Στις νομοθετήσεις για την καινοτομία και την εξυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας, οι προτάσεις νομοθετικές για τη μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής και της πολιτικής ε, αγροτικής ανάπτυξης μετά το 2013 και της ε, ανάπτυξης ε, που, της οποίας ηγείται η τοπική κοινωνία η Επιτροπή των Περιφερειών ζήτησε αύξηση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη, που, ο οποίος έχει πέσει στο 12%. Η αύξηση λοιπόν αυτού του προπολογισμού θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για την κοινωνική ένταξη, τη μείωση τη φτώχεια και τα μέτρα οικονομική ανάπτυξη στι αγροτικέ περιοχέ. Αυτή τη στιγμή, όπω είπα, λαμβάνουν μόνο το 15% του προπολογισμού. Εάν λοιπόν η Γεωργία πρέπει να, εάν η Γεωργία θέλουμε να είναι ανταγωνιστική και πολυλειτουργική, θα πρέπει να δοθεί σημασία στην διαφοροποίηση. Διότι όταν έχουμε μια πολυλειτουργική γεωργία, αυτό συμβάλλει στην αγροτική ανάπτυξη, αλλά δεν αρκεί από μόνο του. Πρέπει και οι άλλοι κοινωνικο-επαγγελματικοί τομεί να κινητοποιηθούν για να προωθήσουν τη βιώσιμη, διαφοροποιημένη και ισορροπημένη ανάπτυξη της των αγροτικών κοινωνιών. Περισσότερη υποστήριξη επίσης πρέπει να δώσει στην τοπική ανάπτυξη. Μόνο το 5% του προϋπολογισμού δίνεται στα leader. Και αυτό δεν αρκεί για να προωθηθούν οι επενδύσεις στις αγροτικές περιοχές στις οποίες επιστρέφει ο κόσμος, ο οποίος ζούσε στις αστικές περιοχές και θέλει τώρα να μειώσει τα έξοδά του και να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης δημιουργώντας δικές του επιχειρήσεις. Δυστυχώς ε, τα άλλα διαρθρωτικά ταμεία επιδεινώνουν περαιτέρω τις, ε, αυτές τις διαφορές. Η μελέτη της ε, Επιτροπής των Περιφερειών που έχετε και εσείς στη διάθεσή σας για τους προϋπολογισμούς που δαπανώνται για την αγροτική ανάπτυξη δείχνει ότι τα ποσά που δίνονται στις ε, αγροτικές περιοχές της Ευρώπης ε, δεν είναι αρκετά. Και η κατάσταση είναι πολύ πιο ανησυχητική σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, διότι τότε είχαμε 32,6% του προϋπολογισμού των διαφθορτικών ταμείων για τις αγροτικές περιοχές, δηλαδή για την περίοδο 2007-2013. Στην τρέχουσα όμως περίοδο το νούμερο είναι μόλις 21,3%. Και αυτό είναι μεγάλη απώλεια για τις γεωργικές περιοχές. Η μείωση στις δαπάνες ε, κυρίως οφείλεται στις περικοπές της χρηματοδότησης που αφιερώνεται στις αγροτικές περιοχές από το Ευρωπαϊκό Ταμείο, ε, το ΕΤΠΑ. Οι αρχικές εκτιμήσεις της DG Regio δείχνουν ότι οι δαπάνες για τις αγροτικές περιοχές έχουν μειωθεί από το 25,8% στην περίοδο 2007-2013 στο, μόλις στο 11,5% στην τρέχουσα περίοδος. Αποτέλεσμα, χρειάζεται αναδρομολόγηση των κονδυλίων. Το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης πρέπει να συμπληρώνει το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο για την Αγροτική Ανάπτυξη, όπως λέει και η Ευρωπαϊκή Συνθήκη, για να μπορέσουμε να έχουμε την εδαφική συνοχή. Όπως είπε και ο κύριος Μπιουκάναν, χρειάζεται άμεση δράση για να έχουμε και καλύτερη επαγγελματική εκπαίδευση στις αγροτικές περιοχές. Μόλις 9% του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου δαπανάτο στις αγροτικές περιοχές στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο και τώρα ο προϋπολογισμός έχει μειωθεί στο 7% για την περίοδο 2014-2020. Ένα νούμερο που μόλις αρκεί για τις βασικές ανάγκες αυτές τις περιοχές και για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αγροτικής εξόδου και της γύρανσης του αγροτικού πληθυσμού. Αυτά πρέπει να ληφθούν υπόψη όσο το δυνατόν στην ενδιάμεση αναθεώρηση του πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου και στην προγραμματική περίοδο μετά το 2020. Συνεχίζω τώρα στο δεύτερο σημείο που είναι η ενσωμάτωση της διάστασης της αγροτικής πολιτικής σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ανάγκες των αγροτικών περιοχών πηγαίνουν πέρα από αυτό που μπορεί να πετύχει η πολιτική ε, γεωργικής ανάπτυξης και έχει λήψεις και σε επίπεδο ποιότητας και ποσότητας. Όλες οι διαρθρωτικές πολιτικές θα πρέπει να έχουν ως βασικό στόχο την αγροτική ανάπτυξη σύμφωνα με το στόχο της εδαφικής συνοχής ε, της συνθήκης της Λισαβόνας. Μία από τις βασικές προτεραιότητες θα πρέπει να είναι η πρόσβαση στα ευρυζωνικά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ένας βασικός παράγοντας ανταγωνισμού και οικονομικής ανάπτυξης. Το 2013 μόλις 25,1% των αγροτικών περιοχών είχαν κάλυψη ευρυζωνική, έναντι 68,1% στις αστικές περιοχές. Παρόλο που η αλληλεξάρτηση μεταξύ αστικών και γεωργικών περιοχών θεωρείται ένας βασικός παράγοντας που πρέπει να εξεταστεί, δεν υπάρχει κάποια πολιτική που να καλύπτει το σημείο αυτό. Έχουμε μόλις ε, μόνο τομεακές προσεγγίσεις από τις ε, Γενικές Διευθύνσεις της Κομισιόν, κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί το ταχύτερο δυνατόν. Είναι σημαντικό λοιπόν να ε, διαφοροποιήσουμε τα σημεία εισόδου και να θέσουμε τη διάσταση της γεωργικής πολιτικής ως ένα συστατικό στοιχείο όλων των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως γίνεται με τις αστικές περιοχές. Θα είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν διάφορα προσκόμματα που σχετίζονται με το εύρος των project, με προκαταλήψεις, αλλά θα ανοίξει ο δρόμος για καλύτερη διασύνδεση και ενσωμάτωση και αλληλεπίδραση μεταξύ αστικών και μη αστικών ε, περιοχών και μέτρων για αυτές τις περιοχές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μία προσέγγιση που να βασίζεται στην τοποθεσία στα επιχειρησιακά προγράμματα. Πέρα από τα πόρου του προπολογισμού, αυτή η προσέγγιση περιμένει, παραμένει περιφερειακή στα, περιφερειακό στοιχείο των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει μεγαλύτερη ε, ευαισθητοποίηση για να έχουμε καλύτερη πολιτική συνοχή και να φτάσουμε καλύτερα στους στόχους της ε, Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Παρόλο λοιπόν που το κοινό στρατηγικό πλαίσιο και οι συμβάσει εταιρική σχέση δημιουργούν ένα υγιέ περιβάλλον για συντονισμό και ολοκλήρωση, θα πρέπει να δούμε ε, τις βασικές καινοτομίες που θα ενισχύσουν την βιωσιμότητα και στην αγροτική ανάπτυξη. Θα πρέπει να έχουμε ανάπτυξη με βάση την τοπική κοινωνία, να έχουμε επενδύσεις σε πράγματα που βρίσκονται στο, κοινό, ε, στο κανονισμό κοινών διατάξεων. Χρειάζονται οι συνέργειες μεταξύ των διαφθορτικών ταμείων επιπλέον. Θα πρέπει να υπάρχουν ε, συγκεκριμένες αρχές που θα εφαρμοστούν. Τέλος, ο σχεδιασμός και εφαρμογή σωστών στρατηγικών που βασίζονται στην ολοκληρωμένη εδαφική προσέγγιση καλεί για περισσότερες, ε, περισσότερους ανθρώπινους πόρους στις αγροτικές περιοχές που έχουν τα μεγαλύτερα προβλήματα. Η Επιτροπή των Περιφερειών επέμεινε σε αυτό το θέμα ε, ως ένα σημαντικό στοιχείο που θα βοηθήσει να, τους ντόπιου ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν και να εφαρμόσουν τις τοπικές, για, τις, για τις τοπικές στρατηγικές και για την εφαρμογή τους. Συμπερασματικά, πριν από 20 χρόνια είχαμε την έγκριση της πρώτης δήλωσης του ΚΟΡΚ στις 9 Νοεμβρίου του 1996 τότε ζητήθηκε μια πιο δίκαιη ισορροπία μεταξύ των αστικών και μη αστικών περιοχών στις δημόσιε δαπάνε και τι επενδύσει σε υποδομέ. Δυστυχώ πρέπει να, να αποδεχτούμε ότι αυτό δεν συμβαίνει σήμερα. Το αντίθετο. Αν θέλουμε να αποφύγουμε μια δεύτερη δήλωση ΚΟΡΚ, την ΚΟΡΚ 2, η οποία έχει εγκριθεί ήδη στις 6 Σεπτεμβρίου 2016, ε, αν θέλουμε να εμποδίσουμε αυτή να παραμείνει απλή, απλά λόγια, πρέπει να φτάσουμε σε ένα επίπεδο rural proofing. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να εξετάζουμε τις μακροοικονομικές και τομεακές πολιτικές από την άποψη της αγροτικής ανάπτυξης. Είναι σημαντικό λοιπόν για να ε, μπορέσουμε να ανδρώσουμε τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα με τέτοιο τρόπο ώστε να φτιάχνουν ναι, λευκές βίβλους ε, για την αγροτική ανάπτυξη που να αποτελούν ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Γι' αυτό ήρθα εδώ σήμερα, για να ζητήσω τη δική σας υποστήριξη για τη δημοσίευση μιας λευκής βίβλου για την αγροτικότητα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για το περιεχόμενο και την ευκρίνεια των λόγων σας. Σημαντική αποστολή μπροστά μας. Έχω τη χαρά να υποδεχτώ τον πρόεδρο Σικώσχη που μου ζητά να συνεχίσω τη διεύθυνση, τη διεξαγωγή των συζητήσεων. Μεγάλη μου χαρά να συντονίζω τις εργασίες μας. Τώρα θα ακούσουμε τους συντονιστές της Επιτροπής ΝΑΤ και τους συντονιστές του Ευρωκοινοβουλίου. Ο κ. Κάστεν Πέτρεσεν έχει το λόγο για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ. Στο πνεύμα της πολιτικής συνοχής που δεν γίνεται σεβαστή, σεβαστό τώρα στην ισορροπία μεταξύ υπαίθρου και πόλεων θα πρέπει να τεθούν οι ώστε η αρχή η βασική να προωθείται. Πρέπει να έχουμε ισορροπία που θα διακρίνει όλες τις πολιτικές επιλογές. Ισότητα δικαιωμάτων για όλους τους πολίτες. Είτε ζουν στην πόλη, είτε ζουν στην Ήπεθρο. Ισοτιμία. Στα μέσα και στις πρακτικές όλων των φορέων. Μεταξύ όλων των περιοχών. Χρειάζεται ανταλλαγή εμπειριών και γνώσεων για να αντιμετωπιστούν οι ιδιωτερότητες της Υπέθρου. Παράδειγμα από τη Δανία. Η Νότια Δανία έχει περιοχές που έχουν προβλήματα οικονομικά. Τι προκλήσει και τα προβλήματα θέλουμε να τα μετατρέψουμε σε δυνατότητε. Οι περιοχές είναι διαφορετικές, διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικά πλεονεκτήματα. Έχουν λιγότερες δυνατότητες όσον αφορά τι ιδιωτικές επιχειρήσεις και ε, παιδεία, εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε όλη τη ζώνη της Νότιας Δανίας. Και αυτό το στηρίζει το Περιφερειακό Φόρουμ. Θέλουμε να συνδυάσουμε πρωτοβουλίε με τι γεωγραφικέ ιδιαιτερότητε κάθε περιοχή. Τριών ειδών πρωτοβουλίε έχουμε. Ένα ειδικό ταμείο για μικρά έργα σε περιοχές της Υπέθρου που συνδέει την Ήπεθρο με περιφερειακά κέντρα και πρωτοβουλίε που εδράζονται επισφαιρικής για τοπική ανάπτυξη έχει υποστηρίξει η περιφέρεια μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή ηλεκτρικού ε, οχηματογωγού και πήραμε χορηγία από τον ορίζοντα 2020 17 εκατομμύρια ευρώ για νέες κατασκευές στην περιοχή. Το πρώτο ηλεκτρικό φέρι θα υλοποιηθεί το 2017. Το χηματογωγό αυτό θα δημιουργήσει θέσει απασχόληση. Και κατά την περίοδο κατασκευή θα δοθεί τεχνογνωσία στο τοπικό ναυπηγείο και θα είναι και μεταφορικό μέσο για ε, του ε, κατοίκου ε, του, νησιού που συνδέεται με την υπηρετική χώρα με αυτό το φέρει. Ευχαριστώ κύριε Πίτερσεν. Ο κ. Ζεμπλεουίξ του ΕΛΚ έχει το λόγο. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, αγαπητή Επιτροπή Γεωργίας, σας απευθύνω θερμό χαιρετισμό και σας ε, μεταφέρω το χαιρετισμό μιας από τις πιο όμορφες ε, περιφέρειες της Πολωνίας, το θα το επιβεβαιώσει και ο πρόεδρος Σικέρσκι και μάλιστα για την περιοχή αυτή η αγροτική ανάπτυξη ε, έχει κομβική σημασία. Σήμερα θα μιλήσω εκ μέρους του ΕΛΚ και εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος θα ήθελα να θίξω δύο θέματα. Το πρώτο αφορά την, ε, τις διακοιμάνσεις ε, των ε, τιμών των γεωργικών προϊόντων. Θεωρούμε ότι η μελλοντική γεωργική πολιτική θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη περιφερειοποιημένων συστημάτων παραγωγής τροφίμων για να ικανοποιήσει την αυξανόμενη ζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, να έχουμε μια απεξαρτοποίηση από την ε, όλο και μεγαλύτερη αστάθεια των παγκόσμιων αγορών πρώτων υλών. Επίσης θα πρέπει να έχουμε διαφοροποίηση των προμηθευτών και να, να τονίσουμε την ανάγκη συνεργασίας με όλους τους κρίκους αλυσίδες και κυρίως να τονίσουμε ε, αλυσίδες βραχίες και ε, να, να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα της αγορές θύλακες, τις ε, αγορές συγκεκριμένων προϊόντων, αλλά να προωθήσουμε και τη βιολογική γεωργία. Αυτά είναι τα βασικά θέματα για τα οποία θα ήθελα σε απευθύνω έκκληση. Ε, Επίσης, ε, το δεύτερο θέμα που με ενδιαφέρει είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στον τομέα του αγροτουρισμού. Ο αγροτουρισμός θα επιλύσει το πρόβλημα της απασχόλησης και της αγροτικής ανάπτυξης για πάρα πολλές περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα ε, ο αγροτουρισμός δεν περιορίζεται μόνο στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά χάρη στη διαφοροποίηση που προσφέρει στηρίζει περισσότερο το βιωτικό επίπεδο των γεωργών. Επίσης ε, συμβάλλει στη διαφύλαξη του γεωργικού τοπίου, του τοπίου της υπαίθρου και προωθεί και τα τοπικά βιοτεχνικά επαγγέλματα. Είναι πολυσχηδής λοιπόν ο, όρος, ρόλος του αγροτουρισμού και γι' αυτό στην ολοκληρωμένη προσέγγιση της ε, μελλοντικής γεωρικής πολιτικής θα πρέπει να στηρίξουμε τον αγροτουρισμό και μάλιστα διασυνοριακές πρωτοβουλίες αγροτουρισμού. Και γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον αγροτουριστικό τομέα και θα τις στηρίξουμε μεταξύ άλλων προσφέροντάς τους ε, βοήθεια στην ε, διαφήμιση και στην προσέλκυση τουριστών και στις αγροτικές ζώνες, στην Ήπεθρο. Επίσης θα πρέπει να βελτιώσουμε την προσβασιμότητα των αγροτικών περιοχών, γιατί γνωρίζουμε ότι από άποψη υποδομών είναι οι πλέον απομονωμένες ε, περιοχές, οι αγροτικές ζώνες. Γι' αυτό θα πρέπει να στηρίξουμε την μεγαλύτερη προσβασιμότητα, τα τοπικά δίκτυα, και φυσικά να ενισχύσουμε τον ψηφιακό τους ε, αλφαβητισμό. Στην δική μας ε, περιφέρεια είχαμε περίπου 1.300 πρωτοβουλίες υπέρ του τοπικού αγροτουρισμού ε, που χρηματοδοτήθηκαν χάρη στα κονδύλια του Ταμείου Ανάπτυξης της Υπέθρου. Και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κάτι διαδικαστικό παρακαλώ τους ομιλητές που θα ακολουθήσουν να προσπαθήσουν να σεβαστούν το χρόνο στη διάθεσή τους, δηλαδή το δίλεπτο που σας διατίθεται. Ξέρω ότι είναι απογοητευτικό και περιοριστικό αυτό. Αλλά ξέρετε ποιοι είναι οι κανόνες για τη διαχείριση του χρόνου εδώ. Ευχαριστώ εκ των προτέρων και δίνω το λόγο στον κύριο Μαρτικάινεν. Uh, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να ελέγξω πρώτα αν μπορώ να μιλήσω ε, φιλανδικά, θα μου πούνε οι διερμηνείς. No, jatkan kuitenkin suomeksi, kun uskon, että tulkkaus φαίνεται Φαίνεται ότι υπάρχουν διερμηνείς που μπορούν να κάνουν διερμηνία των ε, φιλανδικών. Γι' αυτό το λόγο θα ήθελα να αναφερθώ σε κάποια ζητήματα τα οποία θεωρώ σημαντικά. Δεν υπάρχει διερμηνία, οπότε θα συνεχίσω στα αγγλικά. η ε, κατάσταση στις ε, πιο απομακρυσμένες περιοχές μειώνεται. Για ε, κάποιους γεωργούς ε, είναι αδύνατο να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Ε, το εργατικό δυναμικό αλλά και οι ίδιοι κάτοικοι εξαφανίζονται από αυτές τις περιοχές και ύστερα από το 2020 θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες ούτως ώστε να κρατήσουν ζωντανές τις συγκεκριμένες περιοχές. Επίσης, θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών μέσω των ε, δηλώσεων της ε, ύστερα από τις αποφάσεις για τις ποσοστώσεις γάλακτος ε, θα πρέπει να συνεχίσει την, τον διάλογο σχετικά με τη χρήση νέων πρακτικών και την εξέβρεση νέων πρακτικών αλλά και νέες βιώσιμες βάσεις για την γεωργία για να μπορέσει να βελτιωθεί πανευρωπαϊκά και εδώ βέβαια χρειαζόμαστε ε, προσπάθειες με νέα εργαλεία. Ε, τώρα σε αυτό το ε, πλαίσιο έχουμε την συνεδρίαση Food West εδώ πέρα και ήδη από πέρσι είχαμε μία γνωμοδότηση από την ε, δική μου ομάδα θέλουμε βέβαια να έχουμε κάποια ε, αποτελέσματα όμως ε, υπάρχουν μεγάλα, μεγάλες ποσότητες απορριμμάτων τα οποία θα θέλαμε να περιορίσουμε. Σας ευχαριστώ κύριε Μαρτικάινεν. Ο κύριος Στένσον. Thank you, Mr. Chairman. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εκ μέρους ε, της ε, European Alliance ε, θα ήθελα να επαναλάβω ε, κάποια πράγματα. Ε, κατάγομαι από ένα ιδιαίτερα αγροτικό μέρος της Ιρλανδίας. Δεν έχουμε σχεδόν καθόλου broadband σύνθεση. Είχαμε υποσχέσεις από το Κοινοβούλιο και από ε, την Ιρλανδική κυβέρνηση ότι θα έχουμε ε, τέτοια σύνδεση broadband, όμως κάτι τέτοιο δεν συνέβη και θα θέλουμε γι' αυτό να αντιμετωπιστεί άμεσα θέλουμε πρόσβαση ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να ζουν ε, και να εργάζονται στην Δυτική Ιρλανδία. Είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Κατά τη γνώμη μου επικεντρωνόμαστε πάρα πολύ ε, στις αστικές περιοχές ε, και αυτό εις βάρος των αγροτικών περιοχών. Θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό διότι δεν μπορούμε να αστικοποιήσουμε όλε τι περιοχέ, θα πρέπει να κρατήσουμε ζωντανέ και τι αγροτικέ μα περιοχέ. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει ε, να ε, έρθει σε συζήτηση με αυτές τις περιοχές. Λόγω της μείωση των πληθυσμών, πολλά χωριά και μικρέ πόλεις στην Ιρλανδία, αλλά φαντάζομαι και σε όλη την Ευρώπη, δεν έχουν, τις, ε, την δεν έχουν βασικές εγκαταστάσεις. για παράδειγμα ούτε καν αστυνομικά τμήματα και αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Νομίζω ότι στο πρόγραμμα LEADER είναι ιδανικό για να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα και επίσης όσον αφορά την Κομισιόν θα νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις, προ... Ε, ε, προσπάθειές μας ε, να βελτιώσουμε την κακή γη. Θα πρέπει να κρατήσουμε την καλή γη ούτω ώστε οι νέοι να μπορούν να συνεχίσουν να εργάζονται εκεί. Καλωσορίζω την δήλωση ΚΟΡΚ 2 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών μπορούν να αποτελέσουν μέλο, μέρος αυτού και να δώσουν μια νέα ευκαιρία στις αγροτικές περιοχές. Σας παρακαλώ ας μην χαθεί αυτή η ευκαιρία, διότι εμείς ως νομοθέτες και ως πολίτες ε, θα κριθούμε από τα αποτελέσματα σε όλο ε, το ε, ευρωπαϊκό γίγνεσθε το οποίο έχουμε κληρονομήσει. Οπότε ευελπιστώ εν καιρό να μπορέσουμε να το υιοθετήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ κύριε Στένσον. Ο κύριος Άτς έχει το λόγο. you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί Ευρωβουλευτέ. Όπως ακούσατε λέγομαι Arnold Hatch και είμαι μέρος της Επιτροπής Περιφερειών από τη Βόρεια Ιρλανδία επίσημο ηγητή της Επιτροπής των Περιφερειών για την υποστήριξη των νέων αγροτών. Και νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε και ιδιαίτερα η Επιτροπή ότι οι αγροτικές ζώνες είναι πολύ σημαντικές και θα πρέπει να, στηρίξουμε, να τις στηρίξουμε και τις παρούσες αλλά και τις επερχόμενες γενναίες. Και κατά την παρουσίαση ε, τη χθεσινή μου γνωμοδότηση ε, στην Επιτροπή των Περιφερειών για τη στήριξη των νέων ε, αγροτών. Υποστήριξε αυτό το επιχείρημα και μάλιστα έγινε ομόφωνα δεκτή η γνωμοδότησή μου, κάτι που δείχνει τη μεγάλη ομοφωνία και σύμνοια που υπάρχει για αυτό το σημαντικό θέμα. Όπως ξέρετε, μόνο 6% των Ευρωπαίων γεωργών είναι νεότεροι από 35 χρονών. Έχουμε έλλειψη δυστυχώς νέων αγροτών, κάτι που διακυβεύει την οικονομική και κοινωνική βιωσιμότητα των αγροτικών ζωνών. Η προκλήση που αντιμετωπίζει η Ήπεθρος σχετίζεται με τις χαμηλές ε, συγκοινωνίες, χαμηλή βριζονικότητα, στενείς υποδομές μεταφορές και λοιπείς υπηρεσίες παιδείας, υγείας και το καθεξής. Γι' αυτό η στήριξη της γεωργίας είναι προϋπόθεση για την διαφύλαξη της Υπέθρου προκειμένου να υλοποιήσουμε το στόχο Τη ε, εδαφική συνοχή που κατοχυρώνεται στη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και μια και οι νέοι αγρότε είναι οι πιο καινοτόμοι, ε, ειδικά μέτρα του δεύτερου πυλώνα τη ΚΑΠ και επίση ε, τα όρια συνεργασία και προγράμματα τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βελτιώνουμε την κατάσταση, αλλά δεν είναι αρκετά φιλόδοξο όλε αυτέ οι πρωτοβουλίε. Θέλουμε νέους μηχανισμούς και μέτρα για να επιτύχουμε αυτή την ανανέωση των γενεών στη γεωργία και να διαφυλάξουμε την αηφορία της γεωργίας. Γιατί οι χαμηλές αυτές υποδομές είναι τροχοπέδι στην ανάπτυξη και την απασχόληση. Και σίγουρα με τον Brexit θα έχουμε ειδικά προβλήματα και αν δημιουργηθούν σύνορα που θα περικόψουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη και την απασχόλησή μας. Σας ευχαριστούμε κύριε Χάτς. Ολοκληρώσαμε τις παρουσιάσεις των συντονιστών της Επιτροπής των Περιφερειών της Επιτροπής ΝΑΤ και θα ακούσουμε τους συντονιστές της Επιτροπής Γεωργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Αλμπερντές εκ μέρους του ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε συνάδελφοι. Θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι οι αγροτικές περιοχές διαφέρουν μεταξύ των, κρατο... μεταξύ των κρατών μελών. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να προσαρμοστούν αντίστοιχα τα προγράμματα. Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν τις προϋπόθεση διαβίωσης των αστικών περιοχές, διότι εκεί παράγονται τα τρόφιμα, εκεί υπάρχει το νερό. Εμείς είμαστε ε, η ζωή ε, για τις αστικές περιοχές. Η Ευρώπη λοιπόν μπορεί να υποστηρίξει εκεί ούτως ώστε οι αγροτικές περιοχές να λάβουν όθηση. Όμως όχι μονάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και πολιτική κατά τόπους είναι υπεύθυνη. τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα. Ε, εδώ, τα, ε, εδώ και 12 χρόνια ε, εκπροσωπώ τη συγκεκριμένη περιοχή και ήδη από τον ε, πρώτο, ε, πριν από τον Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε ε, στην περιοχή μας υψηλή θνησιμότητα, ε, όμως πλέον είμαστε πολύ καλύτερα. Έχουμε 1,7% ανεργία, τη χαμηλότερη στην ανεργία και για ποιο λόγο συμβαίνει, τη χαμηλότερη στην Γερμανία και για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, διότι έγιναν επενδύσεις και θα πρέπει αυτό ε, να το συζητήσουμε και όσον αφορά το Brown broadband, το οποίο θα πρέπει να γίνει διαθέσιμο, διότι σε περίπτωση που δεν υπήρχε, τότε οι εταιρείε δεν θα μπορούσαν να έρθουν, δεν θα μπορούσαν να έρθουν ε, εταιρείε ε, και να δημιουργηθούν θέσει συνεργασία. Γίνονται επενδύσει στη, στη Βαβαρία πολύ μεγαλύτερε, ύψου 1,5 δι, μεγαλύτερε από ό,τι στην υπόλοιπη Γερμανία και έτσι μπορούν να γίνουν οι προποθέσει ώστε οι αγροτικέ περιοχές να μπορέσουν να επιβιώσουν μελλοντικά και νομίζω ότι θα πρέπει να ε, φροντίσουμε ώστε οι πόροι τη ΝΑΤ να χρησιμοποιηθούν έτσι ώστε να μπορέσουμε ε, να ενισχύσουμε τις περιοχές αυτές θα πρέπει να προσέξουμε πάνω σε αυτό και θα σας παρακαλούσα όσον αφορά τη λευκή Ρίβλα να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας και να εφαρμοστούν όλα αυτά ούτως ώστε να επιτευχθούν στόχοι ανάπτυξης για τις αγροτικές περιοχές. Ευχαριστώ κύριε Ντες. Ο κύριος Δεκάστρο έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ την Επιτροπή των Περιφερειών και ευχαριστώ την Επιτροπή ΝΑΤΑ για τη σημαντική αυτή δυνατότητα που μας δίδεται να πω εμείς ότι υποστηρίζει η ομάδα μου την ανάγκη για μια λευκή βίβλο για την Ήπεθρο και χαιρόμαστε που μπορούμε να υποστηρίξουμε αυτή τη μάχη και όπως είπε και ο συγητής πριν από λίγο είναι μια μάχη που στη διάσκεψη του ΚΟΡΚ αναγνωρίστηκε στην ΚΟΡΚ 2 αναγνώρισε την πολιτική, τις πολιτικές για την άπτυξη της υπαίθρου που θα πρέπει να επεκταθούν οι πολιτικές όχι μόνο προς την αγροτική πολιτική, τη γεωργική πολιτική, αλλά στις πολιτικές της Ένωσης. Μια μεγάλη μάχη είναι αυτή, που είναι μια μάχη που δίδεται κατά της μειοπικής θεωρήσεως των πραγμάτων από τα κάτι μελη Η μεταρρύθμιση της κοινή αγροτικής πολιτικής ολοκληρώθηκε στο Κοινοβούλιο στην προηγούμενη θητεία. Και εκεί αφήσαμε ελεύθερα τα κάτι μέλη να διευρύνουν τις δαπάνες για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Δυστυχώς, όπως υπενθύμιζε ο εισηγητής, λίγες ήταν οι αυξήσεις που δόθηκαν από τα κράτη-μέλη. Μεγάλο κομμάτι των πόρων για την αγροτική πολιτική ε, παρέμειναν στον πρώτο πυλώνα αντί να μεταφερθούν στο δεύτερο. Όπως έλεγε ο εισηγητής, η ΚΑΠ ε, μπορεί μόνη της να ανταποκριθεί σε όλα τα προβλήματα και τις απαιτήσει για μεγαλύτερες προσπάθειες από πλευρά Ευρώπης για πολιτικές αναπτύξεις υπαίθρου. Γι' αυτό είναι σημαντικό να βρούμε νέες λύσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικό να έχουμε τη Λευκή Βίβλο η οποία θα μπορέσει να ερευνήσει και να διευκρινίσει σε ποιο βαθμό οι πολιτικές αυτές μπορούν να βοηθήσουν πλευράς υποδομής στην Ήπεθρο θα μας βοηθήσει να βοηθήσουμε τις κοινότητες και τις περιφέρειες να εφαρμόσουν τις πολιτικές αυτές και να βρουν απαντήσεις στις απαιτήσεις για περισσότερους πόρους. Όπως γνωρίζουμε, η Ευρώπη αυτή μειώνει και δεν αυξάνει τους πόρους. Μειώνονται συνεχώς οι πόροι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ και καλή δουλειά εύχομαι. Ευχαριστώ, κύριε Δικάστρο. Η κυρία Μούλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για αυτή την ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Υπάρχουν πολλές πτυχές της ε, αγροτικής ανάπτυξης που θα πρέπει να υπογραμμιστούν εδώ. Ε, συγκεκριμένα οι μεταφορές, η κίνηση εκπαίδευση με εξειδικευμένα σχολεία στις ε, περιφέρειες. Αυτά πρέπει να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των τοπικών κοινοτήτων. Καλό θα ήταν να έχουμε και άλλες ε, δυνατότητες χρηματοδότησης, ας πούμε από, την, ε, από άλλους τομείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, π.χ. των μεταφορών, έτσι ώστε πολύ στοχοθετημένα να μπορέσουμε να φτάσουμε στο 30, στο ποσοστό αυτό που λέει ότι 30% των γεωργών είναι κάτω των 35 ετών. Θεωρώ ότι καλό θα είναι στο μέλλον να πάρουμε αυτό το σήμα κινδύνου σοβαρά υπόψη μας και να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε πιο ελκυστικές ε, γεωργικές περιοχές για τους νέους. Η κινητικότητα, η, το να ζει κανείς σε μία πόλη και να δουλεύει σε μία άλλη είναι δυνατότητες. Παρόλα αυτά θα πρέπει ε, να ληφθούν υπόψη αυτά τα ζητήματα ε, ταυτόχρονα με θέματα που αφορούν στις εκμεταλλεύσεις, προβλήματα που έχουμε στη Γερμανία και συγκεκριμένα στη Βαβαρία όταν δημιουργούμε δρόμους και όταν δημιουργούνται επιχειρήσεις ε, χάνονται γεωργικές εκτάσεις. Πρέπει λοιπόν να ληφθούν αντισταθμιστικά μέτρα περιβαλλοντικά που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από τον περιβαλλοντικό τομέα και να δοθεί ε, σημασία στην προστασία της βιοποικιλότητας. Νομίζω ότι στη Γερμανία έχουμε πολλά αρνητικά παραδείγματα που καλό θα ήταν να μην τα μιμηθούν άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σένερα τώρα. δεν βλέπω κανένα από την οπότε ο κύριος Λουαζό. Ευχαριστώ. Πολύ λόγο γίνεται στην Επιτροπή Γεωργία σήμερα για την αγροτική ανάπτυξη, αλλά στην πράξη δεν συμβαίνει τίποτα. Πολλά λόγια και ελάχιστα έργα. Έχουμε απερίμωση τη υπαίθρου, κλείσιμο δημοσίων υπηρεσιών, ε, λουκέτα σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ανισότητα μεγάλη ε, και πού οφείλονται όλα αυτά σε μια κοινή γεωργική πολιτική που από το 1992 δεν στηρίζει πια την ευρωπαϊκή γεωργία αλλά επικεντρώνεται περισσότερο στην γεωργοβιομηχανία. Δεν μπορούμε όμως να ζήσουμε χωρίς γεωργία. Και ε, οι περιφέρειες ναι, δεν έχουν περισσότερες εξουσίες, αλλά πρόοδο δεν βλέπουμε. Για παράδειγμα, ε, έχουμε μερικές φορές για τη γεωργία χρηματοδότηση ε, των προγραμμάτων ε, για να προσελκυθούν γιατρούς, αλλά ο αριθμός των φοιτητών στην ιατρική καθορίζεται σε εθνικό επίπεδο. Οπότε σε εθνικό επίπεδο χαράζονται οι πολιτικές και οι περιφέρειες δεν αποφασίζουν για τίποτα, ούτε μπορούν να κάνουν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό. Είμαι από το 2004 σε Δημοτικό Συμβούλιο και ήμουν ε, ε, είμαι ερωτό εδώ και πολλά χρόνια και βλέπω ότι οι σημαντικέ αποφάσει δυστυχώ λαμβάνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ οι περιφέρειες δεν έχουν καμία νομοθετική εξουσία και αρμοδιότητα. Σα ευχαριστώ για την πρόταση Λευκής Βίβλου, που ουσιαστικά όμω επιβεβαιώνει όλες τις προαναφερθήσει μα ανησυχίε δυστυχώ. Ευχαριστώ. Από εδώ και πέρα η διαδικασία που θα ακολουθήσουμε θα είναι εξής. Πρώτα θα δώσω το λόγο στους κυρίους και Λάντς για να σχολιάσουν αυτά που άκουσαν από τους ε, συντονιστές των δύο επιτροπών. Και στο μεταξύ να προετοιμάσουμε το Catch the Eye για τη συζήτηση μετά. Όσοι επιθυμούν το λόγο να το δηλώσουν σηκώνοντα την κάρτα που έχουν μπροστά τους για να μπορέσουμε να καταρτήσουμε ένα κατάλογο αγορητών. Αυτά φυσικά μετά τις δευτερολογίες των κυρίων Μπιουκάναν και Λέντς. Και εφόσον είναι σύμφωνοι. Κύριε Μπιουκάναν, θέλετε το λόγο πρώτα εσείς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευπρόσδεκτα τα σχόλια που ακούσαμε από τους συναδέλφους και από πλευρά Επιτροπής των Περιφερειών και πλευρά Ευρωκοινοβουλίου. Είναι καλό που βλέπουμε ότι έχουμε κοινό όραμα για τη βελτίωση της υπαίθρου. Θέλουμε υποδομές. Θέλουμε να βελτιώσουμε τη δυνατότητα διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου. Είναι ζωτική σημασία σε αυτό. Μην ότι όλοι θα πρέπει να εξετάζουμε την κατάσταση. Να κάνουμε ό,τι μπορούμε για την ανάπτυξη της υπαίθρου. Η, ε, η απομάκρυση των πληθυσμών, η επερήμωση των περιοχών αυτών είναι πρόβλημα. Αν δεν μείνουν οι γεωργοί να καλλιεργούν τη γη, τότε αυτό είναι εις βάρος μας. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε όλα τα μέσα στη διάθεσή μας για να το αποφύγουμε αυτό. Πρέπει να προχωρήσουμε. Είναι υπέροχο που διεξάγεται αυτή η συνεδρίαση. Πολύ καλή ιδέα να δούμε τι μπορεί να γίνει στο μέλλον. Και να αναπτύξουμε δεόντως την ύπεθρο. Θα πρέπει να παράσχουμε υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες αυτό πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προσπαθειών. Ανεξάρτητα από το που διαμένουν, είτε μένουν σε πόλεις, στην Ήπεθρο, είτε στις ακτές. Όλοι οι πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ισότιμα, ανεξαρτήτως τόπου διαμονής. Και θέλουμε έτσι να διαμορφώσουμε τις κοινωνίες που όλοι επιθυμούμε. Ευχαριστώ, κύριε Μπουκάναν. Ο κύριος Λάντς έχει κάποιες απαντήσεις. Ναι, πολύ σύντομα. Κατανοώ ότι συμμεριζόμαστε έναν κοινό στόχο, δηλαδή τη δυνατότητα μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης, ειδικά στις γεωργικές περιοχές. Αναφέραμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γεωργικές περιοχές και συμφωνούμε και με αυτές και σε αυτές. Ας πούμε, τη γέρανση του πληθυσμού, τη μείωση του πληθυσμού, περιβαλλοντικά ζητήματα, την έλλειψη επενδύσεων σε υποδομές, το ζήτημα της ευρυζωνικότητας, που για μένα ως εστονός είναι θέμα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπάρχουν πολλά πράγματα που συμμεριζόμαστε. Όπως ας πούμε η ανάγκη για να υπάρξει μια λευκή βίβλος. Ας αρχίσουμε λοιπόν να εργαζόμαστε επ' αυτού. Αυτό θα είναι το επόμενο βήμα. Μπορούμε όλοι να εργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Λάντς. Πριν περάσουμε στο Catch the Eye και πριν δώσω το λόγο στον επόμενο μιλητή μας, θα ήθελα να χαιρετήσω εγκάρδια τον επόμενο μιλητή, γιατί ήταν από αυτού που έδωσαν μάχη για την Επιτροπή Περιφερειών και μάλιστα ηγήθηκε τη Επιτροπή Περιφερειών για πολλά χρόνια. Και δώσαμε μάχη όχι σε ιδεολογικό επίπεδο, αλλά στην Ήπεθρο ε, με κοινό στόχο την ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών. Τον κύριο Λάγκ, λοιπόν, ε, ευχαριστώ θερμά για τον αγώνα που δίνει υπέρ τη αγροτικότητα. Ε, στο διαμέρισμά του βρέθηκα πριν από λίγο καιρό στη Γαλλία, στη Λοζέρν και εκεί συζητήσαμε εκτενώς τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ορεινή κτηνοτροφία. Έχετε το λόγο κύριε και Ευχαριστώ. Με συγκινείται ιδιαίτερος κύριε Πρόεδρε. Όντως αυτό που είναι κοινό και στους δύο είναι η ισχυρή βούληση να εμφυσίσουμε πνοή ζωής στις αγροτικές ζώνες τα δύο θεσμικά μας όργανα, ε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή των Περιφερειών, με τις αντίστοιχες επιτροπές μας θα πρέπει να κινητοποιηθούν. Και ανησυχώ κάπως βλέποντας το πρόγραμμα ε, και την ατζέντα για τις πόλεις και αντίστοιχα την εξέλιξη των κονδυλίων για την Ήπεθρο. Ε, θα πρέπει λοιπόν να συσπυρώσουμε τις δυνάμεις μας και να δώσουμε από κοινού τον αγώνα υπέρ της Λευκής Βίβλου για τον αγροτικό κόσμο γιατί είχαμε μια πολιτική για τις ορεινές περιοχές και μάλιστα δεν θα με διαψεύσουν μερικοί παρόντες. Ζητήσαμε λοιπόν εκεί ε, την παρουσία της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και χθε ε, στην αρμόδια επιτροπή ε, της Επιτροπής των Περιφερειών έχουμε μεγάλη αστάθεια των γεωργικών τιμών και γι' αυτό έχουμε ένα κοινό διάβημα, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Επιτροπή Περιφερειών ε, δίνοντας έμφαση στις μικρές αλυσίδες διανομής και στην αναβάθμιση της ε, τοπικής παραγωγής, ε, της περιορισμένης σε τοπικές κοινότητες. Και δεν θέλουμε άλλα ψηφιακά χάσματα. Η παραγωγή τεχνολογική εξέλιξη μπορεί να μας επιτρέψει να δώσουμε νέα του και πλεονεκτήματα στις αγροτικές ζώνες, αρκεί να διαμορφώσουμε μια πραγματική αλληλεγγύη και να ε, βρέψουμε από κοινού τους καρπούς ε, των τεχνολογικών εξελίξεων και της ψηφιακής επανάστασης. Χρειαζόμαστε όμως συνεργασία και αλληλεγγύη γι' αυτό και χαίρομαι που η σύμπνοιά μας δείχνει ότι μπορούμε να δώσουμε από κοινού τον αγώνα μας για να διασφαλιστεί η ισορροπία μεταξύ πέθρου και αστικών ζωνών. Γιατί η εδαφική συνοχή αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναπόκειται σε εμάς να κινητοποιηθούμε και να δώσουμε σε αυτό το στόχο στα σάρκα και οστά να τον υλοποιήσουμε για να μην μείνουμε καταδικασμένοι σε μεγάλα αστικά κέντρα αλλά να δώσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση το υπόδειγμα της ισορροπημένης ανάπτυξης των περιφερειών και την, της αγροτικής ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Ροπέ. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους όσους διοργάνωσαν τη συζήτηση. Είναι πολύ σημαντική αυτή η κουβέντα και δεν είναι η πρώτη φορά που διοργανώνουμε αυτού του είδους το διάλογο. Όσοι ακούν όμως τις ε, ομιλίες θα πρέπει να συναγάγουν συμπεράσματα. Εγώ γεννήθηκα στην Ήπεθρο και έζησα επί μακρόν στην Ήπεθρο. Γι' αυτό χαίρομαι που συζητούμε τα προβλήματα που αφορούν την Ήπεθρο. Συζητούμε, αλλά δεν περνάμε πάντα στις λύσεις. Ούτε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά ούτε και σε εθνικό. Όσον αφορά τον άγνωστο παράγοντα για τις τιμές, το μέλλον, τα συστήματα στήριξης, για όλους αυτούς τους λόγους είναι πολύ δύσκολο οι νέοι να αποφασίσουν να μείνουν στην Ήπεθρο. Υπάρχουν πολλοί άγνωστοι παράγοντες. Στον φορά τις βαλτικές χώρες, πρέπει να αναφέρουμε τις διαφορές εισοδημάτων. Είναι πολύ πιο μεγάλα τα εισοδήματα στις πόλεις από ό,τι στην Ήπεθρο. Μια μισή φορά μεγαλύτερο είναι το εισόδημα κάποιου που εργάζεται στην πόλη από ό,τι στην Ήπεθρο. Θα πρέπει λοιπόν να αναφέρουμε τις διαφορές που υπάρχουν όχι μόνο εντός της ίδιας χώρας, αλλά θα πρέπει να αναφέρουμε και τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ κρατών μελών. Γι' αυτό ο κόσμος έχει την τάση να μεταναστεύει. Οι Λιθουανοί βγάζουν πολύ λιγότερα στη Λιθουανία από ό,τι στην Βρετανία ή από ό,τι στη Γερμανία. Αν πάνε να εργαστούν εκεί δηλαδή. Είναι αρκετά αρνητικό το φαινόμενο και γι' αυτό θα πρέπει να σκεφτούμε και να δούμε πώς μπορούμε να κρατήσουμε τον κόσμο στη χώρα του. Πώς να φροντίσουμε ούτως ώστε οι οικογένειες να μην χωρίζονται. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Έχουμε επίγνωση αυτού. Τα προγράμματα όπως το πρόγραμμα Leader θα μπορούσαν να εφαρμόσουν σημαντικότερα μέτρα θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε τα διαθροτικά ταμεία, τους πόρους του Ταμείου Συνοχής, μαζί με τους πόρους του Ταμείου Leader, για να λύσουμε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Χτες, ο καθηγητής της Ισραήλ, από το Ισραήλ, είπε ότι μένουν στην ύπεθρο οι άνθρωποι, διότι είναι αδύνατον να έχουν πρόσβαση σε κάποιες υπηρεσίες, τηλεφωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες στο διαδίκτυο κλπ. Στη Λιθουανία αναπτύσσεται ε, η ψηφιακή τεχνολογία σε καλό επίπεδο, αλλά δεν παρέχονται οι επαρκείς υπηρεσίες για να μειωθούν οι διαφορές μεταξύ υπαίθρου και πόλεων. Γνωρίζουμε όλοι ότι είναι πιο υγιές και καλύτερο να ζει στην Ήπεθρο αλλά αν υπάρχουν αρκετές υπηρεσίες. Αν τους παράσχουμε περισσότερες υπηρεσίες θα μείνει ο κόσμος. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιάρα έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Βρίσκω ε, πολύ ενδιαφέρουσα τη συζήτηση που κάνετε. Θα ήθελα να πω κάποια πράγματα όμως. Δεν έχουμε μονάχα ε, μία ε, δημογραφική αλλαγή αλλά και ένα δημοκρατικό πρόβλημα θα λέγαμε. Οι μεγαλοπόλεις είναι ε, πιο καλά οργανωμένες ε, με αποτέλεσμα ε, να μιλάμε για καλύτερη δημοκρατία. Εκεί όμως δαπανώνται και οι μεγαλύτεροι πόλεις, της στις πόλεις. Έχουμε δηλαδή ε, περιπτώσεις όπου απέχουν πολύ από την ε, πραγματικότητα. Ε, μιλάμε για ένα χώρο όπου οι άνθρωποι, όσον αφορά την αγροτική περιοχή όπου οι άνθρωποι θα θέλαν να εργάζονται. Θα μπορούσαμε να πούμε συγκεκριμένα και να πούμε ότι δεν υπάρχουν αρκετά χρήματα. Το θεωρώ αναγκαίο όμως οι αγροτικές περιοχές μέσω του δεύτερου πυλώνα να ε, προωθηθούν. Έχουμε μια διαφορετική άποψη για το όλο θέμα από αυτό που θα είχαν οι μεγαλοπόλεις και γι' αυτό το λόγο προειδοποιώ από τη δημιουργία διαφόρων ε, ταμείων ε, και τα οποία θα διοικούνται από τις πόλεις. Ένα άλλο ερώτημα το οποίο με απασχολεί είναι ότι έχουμε διάφορα προγράμματα ε, στις αγροτικές περιοχές τα οποία περιλαμβάνουν και τη βάση όπου ε, οι περιφέρειες θα μπορούν να αποφασίζουν από μόνες τους ε, και έχουμε όμως και το πρόβλημα της συγχρηματοδότησης όμως είμαι της άποψης ότι η συγχρηματοδότηση είναι σημαντική αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένα όριο για τις ανοησίες θα μπορούσαμε να πούμε για το 15, για το 20% ε, να υπάρχει ένα ίδιο κεφάλαιο ε, για ε, να δικαιολογεί την, την ύπαρξη των πραγμάτων τα οποία θα μπορούν να εφαρμόζονται από τη βάση. Ρωτάω τους συναδέλφους λοιπόν πώς το βλέπουν αυτό όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Ευχαριστώ με κύριο Γιάρ. Κύριε Γιάρ, ο λόγος του κύριο Εφνίγκ. Ζητώ συγγνώμη που έρχομαι τόσο αργό σε αυτή τη συζήτηση. Φαντάζεστε, φαντάζομαι γνωρίζετε ότι υπήρχε μια κρόαση σε μια άλλη ε, αίθουσα, άρα έπρεπε και εκεί να παραστώ. Θα μιλήσω για το μέλλον της πολιτικής ε, της εμπριζωνικότητας. Ας δούμε λίγο τι συμβαίνει με τη Σκοτία. Εκεί ε, μπαίνει μπροστά, μπαίνουν μπροστά τα τοπικά συμφέροντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δυστυχώ τώρα είναι τεράστια και είναι ιδιαίτερα δύσκολο να προσπαθήσουμε να βρούμε έναν τύπο, μια φόρμουλα που θα είναι ικανή να ικανοποιήσει τους πάντες. Στη Σκοτία θέλουμε περισσότερο να ενδυναμώσουμε τους ντόπιου για να μπορέσουν να έχουν επιδόσεις και να βοηθήσουν στην επιτυχία. Στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχει αυτή η μεικτή εικόνα. Έχουμε τα χωριά τα οποία στο παρελθόν ήταν αγροτικά αλλά τώρα πια έχουν γίνει απλώς εξοχικές κατοικίες. Δεν έχουν κάποια σχέση με τη γεωργία πλέον. Προφανώς όταν δημιουργούνται ευκαιρίες για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις χρειάζεται να δώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες. Νομίζω ότι υπάρχει πραγματική ανάγκη για την αγροτική ανάπτυξη, αλλά πρέπει λίγο να προσέχουμε πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα. Είναι πολύ εύκολο να τα δαπανάμε σε μεγαλεπίβολα σχέδια. Ε, έχουμε όλα αυτά τα χρήματα και πρέπει να δούμε πώς θα τα ξοδέψουμε γιατί δεν μπορούμε πάντοτε να τα ξοδεύουμε όπως θέλουμε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Άγνιο. Αν μου επιτρέπετε θα δώσω το λόγο στον κύριο Σεκέρσκι. Ξέρω ότι και για τον ίδιο είναι πολύ σημαντικό το θέμα της ε, αγροτικής ανάπτυξης. Γι' αυτό θα, δώσω, θα του δώσω το λόγο για να μας πει τις απόψεις του στον τομέα των αρμοδιοτήτων και των ενδιαφερόντων του. Ευχαριστώ. Όπως είπε και ο κύριος Άγνιου, γίνεται παράλληλα η συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων με πολύ σημαντική συζήτηση για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας και πολλοί από τους συναδέλφους της Επιτροπής Γεωργίας ε, παρακολουθούν τη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων. Η δραστηριότητα της Επιτροπής ε, Περιφερειών για την ε, ανάπτυξη πέθρου και την ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών είναι πολύ πλούσιες και γνωστές και συμφωνούμε υπέρ της ανάγκης ολοκληρωμένης προσέγγισης της αγροτικής ανάπτυξης. Δυστυχώς ε, δεν πετυχαίνουμε πάντα αυτή την ολοκληρωμένη προσέγγιση εδώ στον Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πολλοί πιστεύουν ότι ο δεύτερος πυλώνας της κοινή γεωργικής πολιτικής ε, επιλύει τα προβλήματα των αγροτικών περιοχών. Στην πράξη όμως και εξαιτία των εθνικών γεωργικών επιλογών δεν ε, δεν ε, υποστηρίζεται αρκετά η αγροτική ανάπτυξη. Πηγαίνουν κάποια κονδύλια στις επενδύσεις, ε, γίνεται η στήριξη της μεταποιητική βιομηχανίας, αλλά δυστυχώ ελάχιστα κονδύλια από το δεύτερο πυλόν αφιερώνονται στην πραγματική αγροτική ανάπτυξη. Ακόμη και στα, προγράμματα τα αγροπεριβαλλοντικά. Και αναφέρεται βέβαια συχνά η πολιτική συνοχής και στην πολιτική συνοχή έχουμε τα περιφερειακά προγράμματα που σε μεγαλύτερο βαθμό θα έπρεπε να χρηματοδοτούν την αγροτική ανάπτυξη. Βέβαια, όταν ε, λέμε για τα περιφερειακά προγράμματα μας λένε ότι υπάρχει ειδικό πυλώνας, ο δεύτερος. Και γι' αυτό υπάρχουν μεγάλες διαφορές αναπτυξιακές μεταξύ των αγροτικών ζωνών. Γιατί δεν γίνονται δυστυχώς οι ιδέουσες επενδύσεις στις αγροτικές ζώνες και στην Ήπεθρο. Το υπαριθμό είναι ένα πρόβλημα. Είναι το πρόβλημα της ανεργίας. Δεν υπάρχουν αρκετές θέσεις απασχόλησης στην Ήπεθρο. Γι' αυτό και τονίζουμε την ανάγκη της πολυλειτουργικότητας των αγροτικών περιοχών. Και η ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία υποδομών είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να φτιάξουμε τις υποδομές, αλλά οι υποδομές στις αγροτικές ε, περιοχές είναι ακόμη πιο δαπανηρές. Και έτσι τα περισσότερα κονδύλια πηγαίνουν περισσότερο στις αστικές περιοχές και σε επενδύσεις στις αστικές περιοχές, εξού και στη φιλία. Ο περισσότερος κόσμος διαλέγει τις πόλεις για να εγκατασταθεί ως μόνιμο χώρο διαμονής και όχι την Ήπεθρο. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να τονίσουμε την ανάγκη υλοποίηση του στόχου της εδαφικής συνοχής για να μην υπάρχουν πια τόσες διαφορές μεταξύ των περιφερειών και να μην χρειάζεται ο κόσμος να εγκαταλείπει τα χωριά και την ύπεθρο. Και μάλιστα να φροντίσουμε, να δώσουμε κίνητρα ώστε ο κόσμος να επιστρέψει και πάλι στην ύπεθρο και να μην ερημώνονται τα χωριά μας. Αυτό όμως είναι μια αρκετά δαπανηρή επίσης διαδικασία. Θα πρέπει να δημιουργηθούν όλες οι προϋποθέσεις για να καταστεί ελκυστική η ύπεθρος. Είχαμε τις δύο διακηρύξεις την πρώτη και τη δεύτερη διακήρυξη του ΚΟΡΚ τους χωρίζει μία εικοσαετία αλλά έχουν πολύ σημαντικές προτάσεις αυτές οι δύο διακήρυξεις για την ε, ανάπτυξη των αγροτικών ζωνών και πολλές προτάσεις για την καινοτομία και τον εξυγχρονισμό των αγροτικών ζωνών γι' αυτό είναι και είναι πολύ σημαντικές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που δώσατε αυτή τη σφαιρική διάσταση στο θέμα. Ευχαριστώ τους διάφορους που πήραν το λόγο. Ο κ. Μπουκάναν, τον αντιπρόεδρος, ο κ. Λάνς ήταν ο κ. εισηγητής. Ευχαριστώ όλους για το περιεχόμενο των παρεμβάσεών σας, την ευφυΐα των όσων είπατε, δείξατε πόσο ενδιαφέρον το θέμα αυτό της αναπτύξεως υπαίθρου. Κάτι που μας ανησυχεί. Το είπαν πολλοί από σας. Όταν τα μέσα και οι πόροι μειώθηκαν. Ήγηκε η ώρα να έρθει η περίοδος των παχιών αγελάδων. Πρέπει να προβληματιστούμε λοιπόν, να δούμε ποια είναι η σχέση μεταξύ της τοπικής διάστασης με τη γενικότερη, τη σφαιρική. Είναι εξίσου σημαντικό αυτό. Αυτή η κατάσταση μας υποχρεώνει να κινηθούμε σε αυτή την προσέγγιση. Θα πρέπει να εφαρμόσουμε τα όσα σκεφτόμαστε. Πρέπει να μορφωθεί η πολιτική μετά το 2020 και γι' αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε το θέμα της αγροτικότητας, με τη γεωργία. Να λάβουμε υπόψη τα θέματα της διατροφής, της ασφάλειας, ε, του φοδιασμού, τη διατροφή. Αν θέλουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που δημιουργούνται από το περιβάλλον και το κλίμα, εγώ πιστεύω ότι το, η πρόκληση της εδαφικότητας ε, δημιουργείται και είναι πολύ σημαντικό. Θέλουμε να δούμε αν θέλουμε ή δεν θέλουμε ύπεθρο που ζει. Είναι μεγάλος ο κίνδυνος. Το αναφέρατε στις παρεμβάσεις σας αυτό. Και το θέμα της Λευκής Βίβλου το θέσατε. Και η διακομματική η ομάδα Ρούμρα ασχολείται με το θέμα. Η Λευκή Βίβλος είναι πάρα πολύ σημαντική. Στο περιεχόμενο αυτής θα πρέπει συλλογικά να επανατοποθετήσουμε το θέμα της αγροτικότητας σαν μεγάλο διακύβευμα της μελλοντική πολιτικής. Ολοκληρωμένη ανάπτυξη, ολοκληρωμένη ε, ύπεθρος, κινητοποίηση των φορέων, τοπικά προγράμματα, όλα αυτά πρέπει να πάρουν μια διάσταση ούτως ώστε συλλογικά να απαντήσουμε στα μελλοντικά προβλήματα. Το είπατε αυτό, το θέμα των υπηρεσιών, της κινητικότητας, το θέμα της επικοινωνίας. Όλες αυτές οι καινοτομίες θα μας επιτρέψουν να δώσουμε απαντήσεις στα προβλήματα της υπαίθρου και λαμβάνοντας υπόψη και την ποικιλομορφία της υπαίθρου. Θέλουμε να αναμίξουμε δραστηριότητε, θέλουμε να κινηθούμε διαφορετικά. Αυτά πρέπει να απαντηθούν, να δώσει προπτικές η Λευκή Βίβλος προς εξέταση το Ευρωκοινοβούλιο με την Επιτροπή των Περιφερειών, τα δίκτυα, οι διακομματικές ομάδες που ασχολούνται με το θέμα της αγροτικότητας και της υπαίθρου βλέπουν πόσο περίπλοκο είναι το θέμα. Μετά το ΚΟΡΚ 1, στο οποίο είχα τιμή να συμμετάσχω, και στο ΚΟΡΚ 2, ε, και το ΚΟΡΚ 2 είναι πολύ επίκαιρο. Από κοινού πρέπει να απαντήσουμε στα προβλήματα. Αν χρειαστεί να επαναπροσανατολίσουμε και τους πυλώνες ενδεχομένως της κοινή αγροτικής πολιτικής. Το θέμα της υπαίθρου είναι τεράστιο πολιτικό θέμα. Μπορούμε να βασιστούμε σε κοινή συνεργασία. Μπορούμε να τροφοδοτήσουμε και τον προβληματισμό των Επιτροπών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στους επόμενους μήνες και τα χρόνια. Ευχαριστώ για τον πλούτο των όσων είπατε και για τη συλλογική προσπάθεια που δεσμευτήκαμε να καταβάλουμε για να προωθήσουμε την Ήπεθρο. Ευχαριστώ όλους και καλή συνέχεια στις εργασίες σας. Σας εύχομαι. Μάλιστα. μα έμεινε μισή ώρα μέχρι την επόμενη συνεδρίαση, οπότε αν θέλει κανείς το λόγο πολύ ευχαριστώ. Αλλιώς θα διακόψουμε μέχρι τις 5, γιατί στις 5 έχουμε μια ιδιαίτερα σημαντική συνάντηση ε, κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών Γεωργίας και Διεθνούς Εμπορίου με θέμα τις εξωτερικές διαστάσεις των εμπορικών συμφωνιών και τις επιπτώσεις τους ε, στη γεωργία και στην κατάσταση των γεωργών. Και μάλιστα θα έχουμε καλεσμένους τους δύο αρμοδίους επιτρόπους, τον Επίτροπο Γεωργίας τον κύριο Χόγκαν και την Επίτροπο Εξωτερικού Εμπορίου, την κυρία Μάνστρομ. Πολύ σημαντική λοιπόν, βαρισίμαντη η κοινή συνεδρία των δύο επιτροπών που θα ξεκινήσει στις 5 η ώρα. Σας προσκαλώ λοιπόν και αν θέλουν οι καλεσμένοι μας για μία ακόμη φορά το λόγο, πολύ ευχαρίστω. Είδε μη, θα συνεχίσουμε στις 5. Σας ευχαριστώ θερμά για την πρωτοβουλία της Επιτροπής Περιφερειών για την ανάπτυξη της ε, αγροτικής, ε, των αγροτικών ζωνών και της υπαίθρου. Και σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπιουκάναν. Ευχαριστώ κύριε Σεκέρσκι. Χαρήκαμε ιδιαίτερως με τη συμμετοχή μας ε, σε αυτήν την κοινή συνάντηση σε αυτή την κοινή συνεδρίαση και νομίζω ότι καλό θα ήταν να συνεχίσουμε τις επαφές και τη συνεργασία προς όφελος όλων και κυρίως της αγροτικής ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ. Και εμείς προσβλέπουμε σε συνέχιση της αγαστής μας συνεργασίας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για αυτή τη συνάντηση, αυτή την κοινή συνεδρίαση, την πρώτη κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών των Δύο Οργάνων. Σας ευχαριστώ. Διάλειμμα μέχρι τις 5.